Ας ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Σημείο 1. Στην ημερήσια διάταξη, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Ω πρόεδρο προτείνω να διαγράψουμε το σημείο 7 που έχει να κάνει με την διερευνητική αποστολή στο νότιο τμήμα της Ιταλίας οι συνάδελφοι έχουν συναντηθεί, ετοιμάζεται το πρόγραμμα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με όλους τους συναδέλφους δηλαδή, οπότε εμπιστευόμαστε τους συναδέλφους για να ολοκληρωθεί η οργάνωση αυτής της διερευνητικής αποστολής στο Ροζάνο. Σημειώστε ότι υπάρχει προσθήκη στην ημερήσια διάταξη. Μετά τις ψηφοφορίες θα Έχουμε μια σύντομη παρουσίαση της Επιτροπής. Κύριε Φόλ, καλώς ήρθατε. Για την ε, επερχόμενη πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Πολιτείε Συνεργασία για την Προστασία των Δεδομένων. Εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Συνεχίζουμε με το σημείο 2 τώρα στην ημερήσια διάταξη που είναι οι ανακοινώσει του Προέδρου. Πρώτον, προτείνω να εγκρίνουμε τον ορισμό, τη σύσταση μάλλον τον συντονισμό, για τον ορισμό των εξής εισηγητών. Ραούλ Ρομέδα, πράσινη, για την ίση μεταχείριση ατόμων ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την ιδεολογία, την ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεύτερον, Λίδια Γιάροκα από το ΕΛΚ. Είναι η επόμενη συγκήτρια για την έκθεση INI όσον αφορά την κατάσταση των Ρώμα στην Ευρώπη. Τρίτο, Άννα Γκόμες από τους σοσιαλιστές πάλι για την έκθεση INI όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ενίσχυση της ασφάλειας από τα χημικά, βιολογικά και ραδιοενεργά και πυρηνικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια άλλη συγκίτρια, κυρία Κίνγκα Γκάλ από, Α, από το ΕΛΚ, από το ΕΛΚ διορθώνει ο πρόεδρος. Η κυρία Άλλη κίνγκα έχουμε από του σοσιαλιστέ. Για γνωμοδότηση όσον αφορά την πρόσβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πέμπτο. Αντιγόνη Παπαδοπούλου από τους σοσιαλιστές τώρα για τη γνωμοδότηση όσον αφορά μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη ε, θεομηνιών και ανθρωπομηνιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφών που οφείλονται στον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται οι συστάσεις αυτές. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο σημείο 3, που είναι η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένε Πολιτείες για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προβλέπεται ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε. Οπότε, προτείνω να κάνουμε το εξή. Όλοι γνωρίζετε ότι σήμερα το πρωί διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να διατηρήσει για την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια το θέμα στην εμερήσια διάταξη όσον αφορά αυτή την ε, πρόταση για συμφωνία. Οπότε εμεί καλούμεθα να υποβάλουμε σύσταση στην Ολομέλεια. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε την παρουσία του κυρίου Φόλ και του κυρίου Μπουνταρέλη την συμφωνία αυτή με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα, μετά από έναν δεύτερο γύρο συζητήσεων, θα ψηφίσουμε την σύσταση της εισηγήτριάς μας, της κυρίας Γιαννίν Χένις Πλάσχαρτ. Γίνονται συζητήσεις, οπότε σας παρακαλώ προσοχή ως προς τα εξής. Προκειμένου να αποφύγουμε τον κίνδυνο να μην υπάρξει τελικά συνοχή τη στιγμή της ψηφοφορίας βάσει της διαδικασίας της σύμφωνης γνώμης, επιτρέπεται μία μόνο ψηφοφορία. Στην περίπτωση της συμφωνίας αυτής Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένες Πολιτείες TFTP, η συγκήτρια μας υπέβαλε ένα σχέδιο σύστασης που προτείνει Θα περιμένουμε για τη σύμφωνη γνώμη. Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει καλά η ψηφοφορία, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν ψηφίσετε ναι στη σύσταση της εισηγήτριας, αυτό σημαίνει ότι απορρίπτεται τη συμφωνία. Αν ψηφίσετε ναι, σημαίνει όχι για τη συμφωνία. Αντίθετα, αν ψηφίσετε όχι, στην πρόταση της εισηγήτριας, στην έκθεση της εισηγήτριας, αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνείτε με τη σύσταση της εισηγήτριας και ότι άρα δηλαδή εγκρίνεται την συμφωνία. Συνεπώς. Ναι, για διαδικαστικό θέλετε το λόγο, για διαδικαστικό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω δύο θέματα εδώ να θίξω παρακαλώ όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθούμε που σίγουρα επηρεάζει την ψηφοφορία και το, την ισχύ της ψηφοφορίας στην οποία θα οδηγηθούμε σε λίγο. Δύο πράγματα θέλω να πω και σας παρακαλώ εσείς να αποφασίσετε για αυτά γιατί έχει πολύ σημασία για την ισχύ των διαδικασιών μας. Το πρώτο θέμα λοιπόν που θέλω να θίξω είναι το θέμα της μετάφρασης των κειμένων. Εμείς έχουμε πάρει την έκθεση αυτή σε μία και μόνο γλώσσα. Ενώ, από ό,τι ξέρω, πρέπει το κείμενο να διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες προκειμένου να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω στο κείμενο και να ψηφίσουμε. Δεύτερον, θέλω να επιστήσω το Η ψηφοφορία και η σημασία της ψηφοφορίας ποια θα είναι. Διότι το κείμενο που έχουμε μπροστά μας μας συστήνει να μην δώσουμε ακόμα τη σύμφωνη γνώμη μας. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν ψηφίσουμε συν, όπως είπατε πολύ σωστά, συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι δεν δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Όσοι από μας θέλουν να εγκρίνουν τη συμφωνία, σήμερα στην ψηφοφορία αυτή δεν έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Γιατί εδώ καλούμεθα να ψηφίσουμε με ναι ή με όχι. Δηλαδή ε, δεν εγκρίνουμε τη συμφωνία ή την εγκρίνουμε. Οπότε εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διαδικασία. Θα ήθελα εσείς να μας εξηγήσετε καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται το κατά πόσο έγκυρη θα είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας μας ή όχι. Σας τα έχω στείλει και γραπτά όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα πρακτικά πριν προχωρήσουμε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλιώς κινδυνεύει να είναι άκυρη η ψηφοφορία μας. Πρόεδρος. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο διαδικαστικό. Λοιπόν, κύριε Μπουσάτελ, ως ήθιστα. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας. Σημειώνουμε τα ερωτηματικά σας όσον αφορά την διαδικασία ψηφοφορίας και όσον αφορά τις μεταφράσεις που δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες. Αλλά είναι θέμα χρονοδιαγράμματος βλέπετε. Μερικές φορές χρειάζεται να ψηφίσουμε κάτω από ειδικέ ε, συνθήκες, εξαρτάται κατά πόσο είναι ουσίας ή όχι. Οπότε ναι, μεν συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να επιταχύνεται η διαδικασία μεταφράσεων έτσι ώστε όλοι οι ευρωβουλευτές να είναι σε θέση να ενημερώνονται στη γλώσσα τους. Να έχουμε όλες τις μεταφράσεις στη γλώσσα του καθενός μας για την ουσία της ψηφοφορίας. Θα περάσουμε στη γραμματεία το μήνυμα αυτό, ώστε η δουλειά να γίνεται σωστά. Βέβαια, αναφερθήκατε και σε ένα δεύτερο διαδικαστικό που έχει να κάνει με, με το αντικείμενο της ψηφοφορίας. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό εγώ σας εξήγησα λεπτομερώς ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν με τη συνθήκη της Λισαβόνας εδώ πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας Πρώτα απ' όλα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εδώ σήμερα, που ψηφίζουμε τις συστάσεις. Και σας είπα ξεκάθαρα ότι οι συστάσεις στην έκθεση, οι συστάσεις της εισηγήτριας λένε η Επιτροπή μας να μην δώσει ακόμα την σύμφωνη γνώμη της στην συμφωνία. Δεν λέω να απορριφθεί, αλλά να μην προχωρήσουμε σήμερα στη σύμφωνη γνώμη. Και αυτό είναι δεσμευτικό απέναντι στη συνέχεια της συμφωνίας. Δηλαδή αναβάλλεται η θέση σε ισχύ της συμφωνίας που θα ήταν τώρα το Φεβρουάριο. Η συμφωνία δηλαδή δεν θα ισχύει. Όμως αυτή δεν είναι και η τελευταία λέξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή θα τη δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Άρα λοιπόν έχουμε μία εβδομάδα ακόμα στη διάθεσή μας. Εμείς εδώ κάνουμε το καθήκον μας. Ψηφίζουμε τις συστάσεις της εισηγήτριας. Οι συστάσεις συστήνουν να μην δώσουμε ακόμα τη σύμφωνη γνώμη. Όσοι λοιπόν ψηφίσουν ναι στην έκθεση που θα ψηφίσουμε, σημαίνει ότι δίνουν αρνητική ψήφο στην συμφωνία. Όσοι ψηφίσουν κατά της έκθεσης των συστάσεων, άρα ψηφίζουν υπέρ της συμφωνίας. Όσον αφορά την ουσία, έχουμε καιρό ξανά και ξανά να συζητήσουμε το περιεχόμενο ξανά και ξανά. όσον αφορά το SWIFT και το πρόγραμμα αυτό παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Έχουμε καιρό να μπούμε σε βάθος επί της ουσίας της υπόθεσης αυτής. Σήμερα τις συστάσεις της συζυγήτριας μόνο ψηφίζουμε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στη γραμματεία για να πει κάτι όσον αφορά το σύστημα μετάφρασης. Παρακαλώ. Έχουμε λάβει την απάντηση από τις υπηρεσίες που μας πρότεινε το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε για την ψηφοφορία αυτή. Η ψηφοφορία αυτή γίνεται δυνάμει των συστάσεων που περιλαμβάνουν κάποια τμήματα τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Οπότε, σύμφωνα με τους κανόνες, αυτό το κομμάτι, αυτό το τμήμα μπορεί να εξαιρεθεί της ψηφοφορίας. Αλλά η συμφωνία υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, η απόφαση που κυρώνει την ε, συμφωνία υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, οπότε αν θέλετε να επιμείνετε σε αυτό το διαδικαστικό για το θέμα των μεταφράσεων, μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία επί της ε, συμφωνίας. Ναι ή όχι. Στην περίπτωση όμως αυτή, η εισηγητρία θα προτείνει να καταψηφίσουμε όποιος θέλει να υποστηρίξει τη συμφωνία θα πρέπει να ψηφίσει ναι. Αλλά έτσι σημαίνει ότι η συμφωνία θα πάει στην Ολομέλεια δείχνοντας ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όχι άλλα τμήματα που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα. Οπότε το θέμα είναι αν θα ακολουθήσουμε τους κανόνες ή όχι. Αν θα ψηφίσουμε δηλαδή δυνάμει των συστάσεων, αν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν την συμφωνία. Οι συντονιστές έχουν να πούν κάτι. Θα ψηφίσουμε την έκθεση. Θα ψηφίσουμε την έκθεση, όχι την ε, συμφωνία. Θα συνεχίσουμε την ψηφορία ως έχει. Παρακαλώ. Θα πρέπει να παραμείνουμε στην διαδικασία ως έχει, Πρόεδρε. Την έχουν εξηγήσει και οι νομικές μας υπηρεσίες και ο κύριος Ντάνστον έχει στείλει email για την εξήγηση της διαδικασίας τα γλωσσικά προβλήματα, εντάξει, τα κατανοώ, αλλά όλοι οι σκιώδεις συμφώνησαν στις αρχές της εβδομάδας ότι θα ψηφίσουμε στα αγγλικά λόγω έλλειψη χρόνου. Λόγω τη εντολής που λάβαμε από την διάσκεψη των Προέδρων, που τη λάβαμε στις 26 Ιανουαρίου. Προφανώ δεν μπορείτε να περιμένετε να ε, υποβάλω έκθεση και να είναι και μεταφρασμένη σε δύο εβδομάδε. Λυπούμε πολύ γι' αυτό, αλλά μπορώ να μπορούμε να ζητήσουμε από τους διερμηνείς να μεταφράζουν στη γλώσσα του καθενός μας τις, ε, τα κομμάτια για τα οποία υπάρχουν αμφιβολίες. Οι σοσιαλιστές πρόεδρε υποστηρίζουν πλήρως την εισηγήτρια, εκτός από το τελευταίο κομμάτι που θα πρέπει να το διαβάσει. Κατά τα λοιπά, τον υποστηρίζουμε πλήρως. Ωραία. Άλλος κανείς? Πρόεδρε, Το θέμα που ανέφερε ο Μπουσουτήλ έχει μία νομική βάση. Και μετά με το τι λυπόθηκε και από την Γενική Γραμματεία, πρέπει να πω ότι εδώ έχουμε μία υπερβολική γραφειοκρατία. Διότι η έλλειψη χρόνου δεν αποτελεί βάσιμο επιχείρημα, ειδικά για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα να μην μπορεί δηλαδή κανείς να διαβάσει την έκθεση στη γλώσσα του. Αν υπάρχει χρόνος και αν υπάρχει και δυνατότητα να αποφύγουμε επιχειρηματολογία του τύπου ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πράξει αλλιώ και δεν ακολουθήσαμε την ομεμότητα και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο κύριος Διαδεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα έγγραφο μπροστά μας πολύ πολύ πολύ σημαντικό το οποίο υποβαθμίστηκε πρόσφατα αναβαθμίστηκε συγγνώμη πρόσφατα και δεν μπόρεσε να συζητηθεί όπως έπρεπε. Έχουμε τη δεύτερη έκθεση του δικαστού Μπρουγιέχ Είναι μία έκθεση που τη γνωρίζουν λίγοι και την αγνοούν οι περισσότεροι. Και αυτή η έκθεση συμπεριλαμβάνει ορισμένα συμπεράσματα τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε και να λάβουμε υπόψη μας. Διότι δεν πρόκειται για ένα ελάσσον ε, ζήτημα το τι λέει δηλαδή ο δικαστής Μπρουγέρ Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ θα πρέπει να εκφραστεί σχετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρχοπ ε, διαδικαστικό. Η διάσκεψη των Προέδρων Πρόεδρε συμφώνησε ότι σήμερα το απόγευμα θα ψηφίσουμε. Εγώ προτείνω να ψηφίσουμε. Η κυρία Ρομέρο. Σόφι Ινβελτ. Yeah. Υπάρχει ένα νομικό θέμα εδώ. Θα ψηφίσουμε για την ε, συμφωνία αντί για την ε, σύσταση του, της εισηγήτριας, λένε κάποιοι. Αλλά αν δεν έχει κυκλοφορήσει η έκθεση σε όλες τις γλώσσες, πρέπει να έχουμε εδώ πέρα μια συμφωνία για να μην έχουμε νομικό κόλλημα στη διαδικασία. Οπότε θα ψηφίσουμε. Το, σημείο, το θέμα είναι τι θα ψηφίσουμε, τη σύσταση ή τη συμφωνία. Α είναι σαφή λοιπόν τα πράγματα. Θέλετε το λόγο? Διαδικαστικό, Ταβάρες το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την έκθεση ήδη έχει εξηγηθεί, έχει μεταφραστεί, το έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε όλοι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν θα ψηφίσουμε την έκθεση. Απ' την άλλη, όλοι ξέρουμε και ποιο είναι το κείμενο της συμφωνίας, οπότε ας ψηφίσουμε την έκθεση. Πρώτα ο Άλβαρο. Ευχαριστώ. Όχι, διαδικαστικό πρόεδρε. Ένα ερώτημα προς τους ασκιώδεις, γιατί η συγγήτρια έχει πει ότι αν ήταν υπέρ το, του να υπάρχει μόνο η, έκθεση στην, στα αγγλικά και υπήρξε συμφωνία ως προς αυτό να υπάρξει στα αγγλικά, επομένως οι σκιώδεις θα αναφερθούν στην, θα αναφέρονται στην ομάδα τους αν, δεν, αν υπήρχαν προβλήματα. Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα και δούλεψε η συγκήτρια πάνω στην έκθεση, θα πρέπει να θίξουμε τώρα το θέμα. Θα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πιο, πιο πριν. Οπότε οι, οι σκιώδεις θα μας πούνε υπήρξαν προβλήματα ή όχι η Σόφη πρώτα. Να, ρωτήσω το, να ζητήσω από το ΕΛΚ να ξανασκεφθεί το αίτημά του. Όλοι ξέρουμε περί τίνος ε, πρόκειται και ας μην ξεχνούμε ότι η συμφωνία μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μόνο στα αγγλικά. Η διαπραγμάτευση από τους υπουργού έγινε μόνο στα αγγλικά. Οπότε ε, το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να λάβει θέση, γιατί οι πολίτες περιμένουν. Όλοι ξέρουμε τι διακυβεύεται εδώ. Είναι τυπικότητα το αν θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας ε, Χένες ή την ε, συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Εγώ βασίζομαι στο ΕΛΚ να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Κύριε Ποσούτιλ, συμφωνείτε? Ναι, Πρόεδρε να διαβεβαιώσω την Σόφη ότι πραγματικά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά, αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας πολύ σοβαρά και προτείνω να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία με τη σύσταση της εισηγήτρια. όπως δηλαδή είχε στην αρχή Βεβαίω με την προπόθεση ότι αυτό θα καταγράφεται σαφώ στα πρακτικά. Ότι δηλαδή έχουμε δηλώσει τι αμφιβολίε μα για την ισχύ τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε, συμπέρασμα, προχωρούμε. Όπως είχαμε πει στην αρχή. Οπότε θα ψηφίσουμε, θα ακούσουμε την ε, εισηγήτρια και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Όχι. Μόνο, μόνο την έκθεση και μετά να ψηφίσουμε. Εντάξει. Η κυρία Ισηγήτρια έχει το λόγο. Δεν θα μακρηγορήσω, Πρόεδρε, γιατί ε, το επεξηγηματικό μου σημείωμα και οι παλαιότερες συζητήσεις... Μήπως πρέπει να βάλετε τα ακουστικά σας για να με ακούτε, γιατί το μικρόφωνο μου ανοιχτό είναι, Πρόεδρε. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, όπως είπα, γιατί το επεξηγηματικό μου σημείωμα τα λέει όλα. Έχω έρθει σε επαφή με πολλούς συναδέλφους συστήνω στην Επιτροπή να αναβάλει την ε, απόδοση σύμφωνη νόμη, γιατί υπάρχουν πολλές νομικές επιφυλάξει για κάποιες βασικές αρχές όπως αυτή της αναλογικότητας. Αυτή η αρχή θεωρούμε ότι παραβιάζεται δυνάμει των όρων της συμφωνίας. Και να τονίσω ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει πρόσβαση στο Κοινοβούλιο για όλες τις ε, σχετικές πληροφορίες και την βιβλιογραφία, ούτε απαντά στο αίτημά μας για την ε, εντολή για διαπραγμάτευση μιας μόνιμης συμφωνίας. Να υπογραμμίσω για όλους τους, ε, τους συναδέλφους, έχουμε, έρθει, έχουμε δεχτεί εκβιασμούς, πιέσεις, αυτή η ε, δεν υπάρχουν όμως νομικές ε, συνέπειες για την επίσημη ε, έγκριση της συμφωνίας, αλλά βλέπουμε τι ακριβώς κάνει το Συμβούλιο και τι προσπαθεί να περάσει για την επόμενη εβδομάδα και την Ολομέλεια. Ελπίζω να συμφωνήσουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν βρίσκεται εδώ απλώς για να σημειώνει τις απόψεις του Συμβουλίου. Είναι γεγονός ότι το Κοινοβούλιο πάντα ήθελε να. Πάντα του ζητούσαν να, κάνουν, να κάνει υπομονή. Ε, έχει χρόνια που κάνουμε υπομονή όμω. Οπότε δεν, δεν μπορούμε πια να ακούμε ψεύτικε υποσχέσει. Θέλουμε σαφεί δεσμεύσει και τι θέλουμε τώρα. Το, η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο του Συμβουλίου και θα πρέπει να δράσει μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία, αλλά μόνο από ορισμένε προποθέσει. Εγώ έχω μεταφέρει τι απόψει αυτέ και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο και στι αρχέ των ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Okay. Thank you. Ευχαριστούμε. Κύριε Χάνης ναι. Σας ευχαριστούμε. Δεν ε, ανοίγει η συζήτηση εκ νέου. Θα ψηφίσουμε, έτσι. Κύριε Ποσούντελ, θέλετε το λόγο. Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία αυτή έχει να κάνει με τις συστάσεις της εισηγήτριας. Τη συμφωνία θα την ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Τώρα ψηφίζουμε τις συστάσεις. Αν ψηφίσετε ναι στις συστάσεις, σημαίνει όχι στη συμφωνία. Αν ψηφίσετε όχι για τις συστάσεις, αυτό συνάδει με ένα ναι στη συμφωνία. 59 κάρτες έχουμε και 55 είναι τα μέλη. Συνεπώς, τέσσερις κάρτες παραπάνω βρίσκονται στα μηχανήματα. Ευχαριστώ. Τώρα είναι εντάξει. Are we all set and ready? Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για την ψηφοφορία. Ναι. Ωραία. Είναι ονομαστική. Ονομαστική. Είναι ονομαστική η ψηφοφορία ονομαστική ψηφοφορία. Συνεπώς, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. No, no, no. Now, no, we are voting nominal. No, it's not nominal. It's nominal. Because I am. Okay. Are we voting? Okay. Are we voted? So we... Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Συνεπώς, ναι, υπέρ της σύστασης, εγκρίνεται η πρόταση της εισηγήτριας. Εντάξει. Okay. Then let's proceed. Καλώς. Επόμενο σημείο. Παρακαλώ, ησυχία λίγο. Movement of Κυκλοφορία προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής. Παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κοέγιο για τη θεώρηση μακράς διαμονής. Εδώ καλύπτονται δύο προτάσεις επιτροπών που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση ισχύ της Λισαβόνας. Οι δύο αυτές προτάσεις έχουν να κάνουν με τη διαδικασία συναπόφασης και αποφασίσαμε να τις συγχωνεύσουμε για να έχουμε μία ενιαία διαδικασία. Υπάρχουν πέντε τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, αλλά μετά αποσύρθηκαν. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υπέβαλε τις νομοδοτήσεις ο εισηγητής με τους ε, σκιώδεις εισηγητές κατέληξαν σε ένα συμβιβαστικό κείμενο προκειμένου να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Το συμβιβαστικό κείμενο εστάλει όλα τα μέλη της Επιτροπής μας ΛΥΜΠΕ με τον κατάλογο ψηφοφοριών και το σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου. Δύο πράγματα θα ψηφίσουμε λοιπόν. Πρώτον, το συμβαστικό κείμενο στο σύνολό του. Η δεύτερη ψηφοφορία έχει να κάνει με το σχέδιο ε, ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου. Εφόσον δεν γίνει δεκτός ο συμβιβασμός στο συμβαστικό κείμενο και πρέπει μετά να ψηφίσουμε κάθε άρθρο χωριστά, ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον εναλλακτικό κατάλογο ψηφοφοριών που εστάλει επίσης χτε στους ευρωβουλευτές της ΛΥΜΠΕ. Οπότε θα δώσουμε το λόγο πρώτα απ' όλα στον εισηγητή, τον κύριο Κοέγιο, και μετά θα ζητήσουμε από την Ισπανική Προεδρία να δει κατά πόσο το συμβαστικό κείμενο που έχει εγκρίνει σήμερα η ΛΥΜΕ μπορεί να πάρει επιβεβαίωση από την Κορεπέρ για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Κύριε Κοέγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε όλους τους σκιώδες εισηγητές θέλω να πω ευχαριστώ πολύ, όπως επίσης και στους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της Ισπανικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία τους για να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα κείμενο με τη βοήθεια των σκιωδών εισηγητών με διάφορες συναντήσεις που είχαμε και όπου λάβαμε υπόψη μας τις διάφορες προτάσεις που έγιναν. Όντω θέλουμε να διασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στον ε, χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άτομα με θεώρηση μακράς διαμονής. Λάβαμε υπόψη μας τις προδιαγραφές για ασφάλεια, λάβαμε υπόψη μας επίσης το θέμα της προστασίας των δεδομένων και το δικαίωμα ενημέρωσης. Νομίζω ότι έχω συμπεριλάβει όλες τις προτάσεις που ακούστηκαν και έτσι έχουμε καταλήξει σε ένα συνενετικό κείμενο, ιδιαίτερα ισορροπημένο. Έπρεπε και πρέπει να φτάσουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση γιατί ισχύουν τώρα νέοι μηχανισμοί νομοθετικοί που αναφέρονται στο δικαίωμα μακράς διαμονής. Οπότε έπρεπε γρήγορα να πάρουμε μια απόφαση αποφεύγοντας να τους έχουμε σαν ομήρους τους ανθρώπους αυτούς που έχουν θεώρηση μακράς διαμονής. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Προεδρίας. Ροντρίγεθ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως ε, εξαιρετικά ανέφερε ο κύριος Κοέλιο, τα τρία θεσμικά όργανα κάναν ό,τι μπορούσαν για να σταματήσουν τα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλησαν να λύσουν και το θέμα της βίζας, της θεώρησης για πολλούς ε, αλλοδαπούς ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς με τον εισηγητή προσπαθούμε να βρούμε ένα συμβιβαστικό κείμενο τις τελευταίες μέρες όπου εξισορροπείται η ελευθερία διακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο χώρο Σέγγεν και ασφάλειας. Υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες βέβαια εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών, μας υποστηρίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη και όταν θα έχουμε την τελική συμφωνία στο Συμβούλιο θα την κοινοποιήσουμε και στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Ροντρίγκε για την Κομισιόν. Η κυρία Νάγκη. Δεν είναι εδώ η κυρία Νάγκη. Δεν θα πάρει κανείς το λόγο. Εντάξει. Οπότε ας ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτα για το συμβιβαστικό κείμενο στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Ωραία. Εγκρίνεται το συμβαστικό κείμενο. Πάμε στη δεύτερη ψηφοφορία για το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται και το σχέδιο ψηφίσματος. Οπότε, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στην, ε, στην σύνοδο του Μαρτίου. Πριν την ψηφοφορία, η Επιτροπή Γιούρη θα πρέπει να εγκρίνει τις αλλαγές στη νομική βάση του σχεδίου κανονισμού λόγω της συγχώνευσης των δύο διαδικασιών. Εγώ έχω στείλει μια επιστολή στην Επιτροπή Γιούρη και έχω ζητήσει την έγκρισή τους. Και με ενημέρωσαν ότι η Επιτροπή Γιούρη μπορεί να λάβει θέση στη Σύνοδο του Μαρτίου στο Στρασβούργο. Now we are opening... Οπότε, ο κύριος Τζόναθαν Φόλ θα έρθει τώρα, Γενικός Διευθυντής από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας κάνει μια παρουσίαση για την ε, συμφωνία που επίκειται για την προστασία των δεδομένων. Κύριε Φόλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Η Επιτροπή και διάφορες ε, προεδρίες ε, συζητούν τις αρχές για την προστασία των δεδομένων με τις αρχές των ΙΠΑ εδώ και καιρό δυνάμει μιας έντολης που έχει δοθεί και ανανεωθεί αρκετές φορές για τις ε, διάφορες προεδρίες και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία μεταξύ ημών και των ε, Αμερικανών να δούμε αν υπάρχουν κοινά στοιχεία στα νομικά μας ε, συστήματα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όντως, Υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία, βεβαίως υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές. Και συζητούμε σε, με διάφορους τρόπους το πώς μια κοινή, μια κοινή δέσμη αρχών θα μπορούσε να τύχει υποστήριξη και από τους δύο. Κάποια θέματα εξακολουθούν να είναι αντιφατικά, οπότε θα τύχουν περαιτέρω συζήτηση. Τώρα όμως που έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρούμε πως μια κοινη μια δεσμη αρχων θα μπορουσε να τυχει υποστηριξη και απο τους δυο καποια θεματα επιτέλους η ώρα να γίνει αυτό σε μια πιο ασφαλή και δεσμευτική βάση, οπότε η Κομισιόν ετοιμάζεται να προτείνει την, την θέση σε ισχύ εντολή για επίσημε διαπραγματεύσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και για την ανταλλαγή δεδομένων και ποιε είναι οι προποθέσει σύμφωνα με τι οποίε θα μπορούσαν να ανταλλάσσονται ε, πληροφορίε, προσωπικά δεδομένα για θέματα νομικά. Θα συμφωνείτε όλοι ότι θα ήταν καλό και σκόπιμο να γίνει ευρεία διαβούλευση, ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό και αυτό ξεκινούμε να κάνουμε τώρα. Πριν έρθουμε δηλαδή εδώ ενώπιόν σας, θα κάνουμε πολλές συζητήσεις και με το Συμβούλιο Θέλουμε όμως να ενθαρρύνουμε την έναρξη μιας συζήτησης για το πώς θα έχει αυτή η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Κομισιόν, δυνάμει και της συνθήκης της Λισαβόνας, θα είναι ο διαπραγματευτής. Αυτή είναι η ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά βεβαίως. Και σε αυτό το, την πρωταρχική φάση θα θέλαμε να ε, εμπλακούμε σε ενεργές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία λοιπόν και στο τέλος της διαδικασίας αυτής η Κομισιόν θα υποβάλει την ε, συμφωνία. Από τώρα όμως μέχρι τότε θα υπάρξουν πολλές δυνατότητες για συζήτηση όλων αυτών των ακανθοδών θεμάτων. Μόλις καταλήξουμε σε συμφωνία, και αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει, μόλις λοιπόν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα θέματα μεμονωμένων ανταλλαγών δεδομένων. Ίσως τα πράγματα τότε να είναι πιο απλά, γιατί ούτως ή άλλως θα υπάρχει και ένα συμπεφωνημένο ε, διατλαντικό πλαίσιο. Ε, δεν θα είναι όμως εύκολο να φτάσουμε εκεί. Οι συζητήσεις και εδώ και για το SWIFT και για το PNR και για άλλα σχετικά θέματα έδειξαν ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα Βέβαια, για κάποιους ε, τομείς ε, ε, με τη ΣΥΠΑ μοιραζόμαστε κάποιες αρχέ και κάποια κοινά νομικά πρότυπα, αλλά τώρα το πώ προστατεύουμε εμείς και αυτοί τα προσωπικά μας δεδομένα είναι τελείως διαφορετικό. Για να καταλήξουμε λοιπόν επί τη βάση αυτή μια, σε κοινή αρχή, σε κοινέ αρχές θα είναι δύσκολο. Το Κοινοβούλιο θα, είναι, θα βοηθήσει την Κομισιόν ως προς το θέμα αυτό. Οι δύο επίτροποι που θα ασχοληθούν με το θέμα έχουν αφοσιωθεί σε αυτό και βεβαίως προσβλέπουμε στι συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Ενφέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο μας ζητάει διατλαντική συμφωνία για την προστασία δεδομένων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι θέλουμε δηλαδή. Οπότε χαιρόμαστε ότι οι ιδέες ακούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως επίσης για πάρα πολύ καιρό το κοινοβούλιο μας ζητάει να συμμετέχει στη διαδικασία. Και πάλι η ελευθερία των πολιτών τυχαίνει μεταχείριση ως να πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία σαν να μην συμμετέχει στι διαπραγματεύσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία που κάναμε πριν από δύο λεπτά πρέπει να αποτελέσει ένα μάθημα για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ναι, θέλουμε συμφωνία, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε σε τέτοια συμφωνία μετά από ανοιχτή συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Να συμμετέχουμε στι διαπραγματεύσει. Υπενθυμίζω λοιπόν στον κύριο Φόλ και του συναδέρφους ότι η κυρία Ρέντινγκ μα ανακοίνωσε αναθεώρηση ολόκληρου του πλαισίου για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία και την συμφωνία πλαίσιο για την προστασία στον τρίτο πυλώνα. Όπως επίσης και κατά τομέα διακανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Ας περιμένουμε λοιπόν να έχουμε τις δικές μας προδιαγραφές πρώτα και σε αυτές να βασιστούμε για να έχουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην βιαστούμε δηλαδή για μια νέα συμφωνία και οδηγηθούμε στην ίδια κατάσταση όπως οδηγηθήκαμε με το SWIFT. Και θα το δούμε και για άλλες διεθνείς συμφωνίες. Επιτέλους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με πλήρη δημοκρατική νομιμότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ινχετφέλτ. Άλλες ερωτήσεις. Καλώς. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στο σημείο 5. ή μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, υπεπιθύσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσου προσανατολισμού. Εδώ συζητάμε την κατάσταση πρόοδου των διαπραγματεύσεων. Θα ακούσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Ραούλ Ρωμέβα πρώτα. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοίμασε γνωμοδότηση για την ίση μεταχείριση. Η προηγούμενη έκθεση Βέγγα εγκρίθηκε στην Ολομέλεια τον Απρίλιο του 2009. Στην προηγούμενη θητεία δηλαδή. Βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης. Τώρα με την συνθήκη της Λισαβόνας, το θέμα αυτό απαιτείται σύμφωνη γνώμη. Το άρθρο 19 της ε, συνθήκης και έτσι ορίστηκε νέος εισηγητής μόλις που είναι ο κύριος Ρωμέβα. Ας δώσουμε το λόγο λοιπόν στον ε, εισηγητή μας και μετά θα ακούσουμε την κυρία Λίν που είναι συγγήτρια που συνεργάζεται με την ΛΥΜΠΕ από την Επιτροπή Απασχόλησης. Σήμερα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πρέπει να πω ότι αυτό που κάνουμε είναι να συνεχίζουμε τη δουλειά που είχε ξεκινήσει η Κατερίνα Μπόιτεμπεργκ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ήταν μια δουλειά πολύ δύσκολη και κατάφερε να ισορροπήσει διαφορετικές ευαισθησίες για ένα θέμα πολύ σημαντικό και πρέπει να σεβαστούμε τη δουλειά που έγινε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση στη συζήτηση που θα γίνει και στην εντολή που θα δοθεί στο Κοινοβούλιο και στον εισηγητή για το διάλογο με το Συμβούλιο ώστε να προχωρήσουμε ε, στην πρόταση, στη συζήτηση της πρότασης της οδηγίας. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω πρώτα είναι να χρησιμοποιήσουμε την προηγούμενη εντολή ως διαπραγματευτική βάση και η συζήτηση που θα έχουμε με το Συμβούλιο στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας να βασιστούν στην προηγούμενη εντολή. Βέβαια εμεί θα ακούσουμε το Συμβούλιο που θα μας εκθέσει την κατάσταση ε, σήμερα στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε ποιοι, συγγνώμη, πού βρίσκονται τα προβλήματα που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε σήμερα. Λοιπόν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορέσουμε να λύσουμε σε αυτή την Προεδρία ή όχι. Ποιες χώρες δημιουργούν εμπόδια και γιατί. Και επειδή είναι εδώ και Κομισιόν, να ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της Κομισιόν σε όλη αυτή τη συζήτηση. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η Κομισιόν σε όλα αυτά εμείς έχουμε μερικά κείμενα, αρχικά κείμενα για να δούμε το πώς εξελίσσεται η συζήτηση στο Συμβούλιο. Δεν είναι το ολοκληρωμένο κείμενο, αλλά θέλουμε να ξέρουμε από άποψη χρονοδιαγράμματος πότε θα το έχουμε για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε στο σύνολό του. Θέλω να επαναλάβω αυτή τη βούληση του Κοινοβουλίου να συνεισφέρει στο διάλογο και να ζητήσει και αυτήν την ε, ρύθμιση του διαλόγου κατά τέτοιο τρόπο που να μας οδηγήσει στην έγκριση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θέλουν να μιλήσουν, ε, το Συμβούλιο και η Κομισιόν θέλουν να μιλήσουν, αλλά και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Μου είπανε ότι η κυρία Λίνη Συγήτρια από την Επιτροπή Επασχόλησης κλήθηκε να έρθει εδώ. Την καλέσαμε. Δεν ξέρω, είναι εδώ. Να πάρει το λόγο. Την έχουμε καλέσει να έρθει. Όχι από ό,τι φαίνεται. Καλά, τι να κάνουμε. Η Ισπανική Προεδρία και η Κομισιόν θα μπορούσαν να πάρουν το λόγο τώρα η κυρία Σέρα από την Ισπανική Προεδρία πρώτα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που με καλέσατε να έρθω εδώ σήμερα και να σας παρουσιάσω λίγο την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία αυτή. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο οδηγίας τον Ιούλιο του 2008. Δεν θα επεκταθώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια που είναι εδώ εκπρόσωπος της Επιτροπής να σας τα πει. Εκείνος θα σας μιλήσει για την πρόταση οδηγίας που υπέβαλαν. Αυτό όμως που θέλω εγώ να ξέρετε είναι ότι πρόκειται για μια οδηγία για την οποία εφαρμόζεται η αρχή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσου προσανατολισμού. Τελικά δηλαδή πρόκειται για μια οδηγία η οποία συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο του σημερινού άρθρου 19, τέος άρθρο 3, ε, 13. Το συμπληρώνει λοιπόν με τις τέσσερις αυτές διαφορετικές διακρίσεις που βρισκόταν σε κρεμότητα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν ήταν έτοιμη 2 Ιουλίου και το Συμβούλιο ξεκίνησε να συζητάει την πρόταση αυτή υπό Γαλλική Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2008 δηλαδή. Η Γαλλική Προεδρία αφιέρωσε στην οδηγία αυτή έξι συνεδριάσεις. Προχωρήσαμε πολύ όσον αφορά τη γνώση του πλαισίου, της οδηγίας κλπ. Και εκεί εντοπίστηκαν πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Είναι δηλαδή μια πολύ σημαντική οδηγία, αλλά συγχρόνως και μια περίπλοκη οδηγία, που ακριβώς γι' αυτό χρειάστηκε χρόνος με διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Η Γαλλική Προεδρία, σας είπα, αφιέρωσε έξι συνεδριάσεις στην οδηγία αυτή. Και επειδή υπήρχαν προβλήματα, αμφιβολίες όσον αφορά κάποιες έννοιες που χρειαζόντουσαν διευκρινήσεις, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου κατέληξε σε γνωμοδότηση εξηγώντας πώς είχε το θέμα της κοινοτικής αρμοδιότητας στο τομέα εφαρμογής των ε, ενιών επικουρικότητα, αναλογικότητα κλπ. Τελικά, Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας υπήρξε ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, όπου οι Υπουργοί εξέφρασαν τις απόψεις τους για την οδηγία αυτή, υπογραμμίζοντας πόσο μεγάλη σημασία έχουν όλοι αυτοί οι τομείς τους οποίους θίγει η οδηγία και είπαν ότι θέλαν διαπραγματεύσεις, μια που υπήρχαν ακόμα αρκετές έννοιες που χρειαζόντουσαν παρετέρω διευκρίνηση, νομική βάση, πεδίο εφαρμογή κλπ. Η Τσέχικη Προεδρία τώρα επίσης έγιναν συνεδριάσεις για την οδηγία αυτή που επικεντρώθηκαν κυρίως στον τομέα της αναπηρίας. Εκεί είχαμε σημαντική πρόοδο. Ιδιαίτερα είχαμε προσέγγιση της πρότασης στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης είχαμε και μια έκθεση πρόοδου υπό Τσεχική Προεδρία. Τελικά, κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης προεδρίας της Σουηδικής, επίσης έγιναν συνεδριάσεις όπου σε επίπεδο Συμβουλίου ξαναείδαν ολόκληρη την οδηγία. Ξεκίνησαν από το άρθρο 1 και προχώρησαν ολόκληρη, σε ολόκληρη την οδηγία κατά την Σουηδική Προεδρία και προχώρησαν πάρα πολύ σε θέματα πιο τεχνικά, σε θέματα ορίων πεδίου εφαρμογή κλπ. Η Σουηδική Προεδρία ετοίμασε επίσης μια έκθεση πρόοδου. στη συνεδρίες του Συμβουλίου Εύσκο του Νοεμβρίου υπογραμμίστηκε η πρόοδος που είχε επιτευχθεί όσον αφορά την οδηγία αυτή υπογραμμίστηκε επίσης και το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία παραμένουν σε κρεμότητα. Η Ισπανική Προεδρία τώρα, που μόλις ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, τώρα τον Ιανουάριο, είχε μια πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Κοινωνικών Υποθέσεων για την οδηγία αυτή στις 22 του μήνα που μας πέρασε. Στόχο τη Προεδρία τη Ισπανική είναι να αφιερώσει την οδηγία αυτή όσο γίνονται περισσότερε προσπάθειες για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει και να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων τον Ιούνιο. Ιουνίου. Αυτή είναι η πρόθεση τη ισπανική προεδρία. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει. Τώρα λιγάκι για να καταλάβετε γιατί είναι περίπλοκη αυτή η οδηγία, όσοι δεν τη γνωρίζετε καλά. Σαν παράδειγμα μόνο θα σας δώσω το εξή. Υπάρχουν σημεία σημαντικά και δύσκολα, που είναι ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων, για παράδειγμα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Νομική βάση που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπα και πριν, είναι το άρθρο 19, το σημερινό άρθρο 19, της ηθίκης της Λισαβόνας, ενώ πριν ήταν το 13. Τα θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας επίσης. Γι' αυτό, και αυτό φαίνεται και σε κάθε συζήτηση που γίνεται, χρειάζεται σαφής ορισμός και διάκριση των αρμοδιοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και χωρών μελών από την άλλη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την παιδεία. Ένα άλλο περίπλοκο σημείο επίσης είναι ό,τι έχει να κάνει με διαφορές μεταχείρισης που επιτρέπει η οδηγία. Με άλλα λόγια δηλαδή, τι εξαιρέσεις βάζουμε στην ίση μεταχείριση των προσώπων. Λέει λοιπόν η οδηγία ότι υπάρχει μία διαφορετική μεταχείριση, λόγω για παράδειγμα, που δεν οφείλεται όμως σε διάκριση. Η διαφορετική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία που δεν έχει να κάνει όμως με διάκριση. Ότι δεν μπορούν τέτοιες συμπεριφορέ να θεωρηθούν διάκριση. Αρκεί ο στόχος της διάκρισης αυτής, της διαφοράς αυτής, να είναι, η λόγοι αυτοί να είναι θεμητοί λοιπόν και αναγκαίοι. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Από την άλλη, δεν είναι εύκολο να πει κανεί από πριν κατά πόσο τα μέσα που χρησιμοποιούνται για διαφορετική μεταχείριση οδηγούν σε διάκριση ή όχι, ανάλογα με το αν είναι αναγκαία ή όχι, την αναγκαία ότι δεν είναι. Υπάρχουν και άλλες έννοιες που εξακολουθούμε να συζητάμε και που πρέπει να διευκρινιστούν παρετέρω, όπως είναι το θέμα της πρόσβασης των ε, λογικών ε, διορθώσεων όταν κάποιος με αναπηρία θέλει να έχει πρόσβαση σε ένα κτίριο και δεν μπορεί γιατί δεν υπάρχουν ε, ράμπες, τι διορθώσεις μπορούν να γίνουν στα κτίρια που να είναι λογικές για να μπορεί το άτομο αυτό να έχει πρόσβαση σε αυτό το κτίριο. Και αυτό είναι πολύ λογικό, αλλά έχει μεγάλη σημασία και εξακολουθούμε να το συζητάμε. Δεν έχει τελειώσει. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι ότι έχει να κάνει με το οικονομικό άχθος. Προσαρμογή κτηρίων όπως λέγαμε, προσαρμογή αρχαιολογικών χώρων για άτομα με αναπηρίες. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να ξεκαθαριστεί πλήρως. Και τα καινούρια κτίρια και αρχαιολογικοί χώροι, τα ιστορικά μνημεία. Οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν, πρέπει να είναι λογικές για να έχουν πρόσβαση και τα άτομα με αναπηρίες. Όλες αυτές λοιπόν είναι έννοιες περίπλοκες, δύσκολες χρειάζονται διευκρίνηση. Όπως ό,τι έχει να κάνει με την διάκριση που δεν είναι πάντα άμεση, υπάρχει και η έμεση διάκριση. Αναφέρεται και σε άλλες οδηγίες. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να τύχει διακριτική μεταχείριση επειδή έχει ένα παιδί με αναπηρίες. Αυτή είναι η έμεση διάκριση ή διάκριση λόγω σφάλματος. Να υπάρξει διάκριση σε βάρος κάποιου ατόμου από λάθος, να νομίζουμε ότι κάτι έχει κάνει που δεν έχει κάνει. Το άλλο θέμα που απασχολεί εδώ είναι και η όχληση. Όλα αυτά είναι παραδείγματα που σας δίνω για να αντιληφθείτε ότι παρόλο που έχουμε πολλούς μήνες που συζητάμε για την οδηγία αυτή, εξακολουθούμε να τη συζητάμε, να τη διορθώνουμε, να την προσαρμόζουμε έτσι ώστε η κατάσταση να είναι ξεκάθαρη και να μην καταλήξει τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίζει για την ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας αυτής. Θέλουμε δηλαδή να είναι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρη για όλους. Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στη συνέχεια. Γίνονται συζητήσεις λοιπόν στο Συμβούλιο ακόμα. Μέσα Φεβρουαρίου έχουμε την επόμενη συνάντηση για αυτή την οδηγία. Και σίγουρα θα φροντίσουμε να γίνουν οι συνεδριάσεις που χρειάζονται ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου επί Ισπανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ κυρία Σιέρα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Όλσον είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Η Προεδρία ήταν εξαντλητική. Κάποια σχόλια όμως θα κάνω κι εγώ. Η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει μέτρα στον τομέα αυτό προέρχεται από την συνθήκη του Άμστερνταμ, το άρθρο 13. Οπότε το Συμβούλιο επί τη βάση αυτή έχει εγκρίνει τρεις οδηγίες. Μία που καλύπτει τον, ε, την ε, απασχόληση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες επί τη βάση ε, διακριτικής μεταχείρισης λόγω προέλευσης. Επίσης, υπάρχει οδηγία για την διακριτική μεταχείριση ανάλογα με το φύλλο και τρίτη οδηγία που καλύπτει τους υπόλοιπους τομείς. Ε, γενετήσιος ε, προσανατολισμός, αναπηρίες κλπ. Αλλά το έχει και ως στόχο τον, την απασχόληση, αλλά όχι τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν και η πολιτική συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτό έχει ως επίκεντρο το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας για διάφορους λόγους. Και η οδηγία αυτή στοχεύει στο να γεμίσει τα κενά που υπάρχουν στην προστασία, να καλύψει δηλαδή τα κενά που υπάρχουν στους διάφορους τομείς, ώστε όλοι οι τομείς να είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο. Το Κοινοβούλιο βέβαια έχει εγκρίνει μια αρκετά πλήρη υποστηρικτική γνωμοδότηση τον Απρίλιο του 2009 και η Κομισιόν και το Συμβούλιο την έχουν μελετήσει και την έχουν συμπεριλάβει στις συζητήσεις με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Η Κομισιόν εξακολουθεί να έχει υπόψη της την έκθεση αυτή όταν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στο Συμβούλιο. Τέλος, Μπορεί να το ανέφερε βέβαια η Προεδρία ή ο εισηγητή, αλλά υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ομοφωνία εδώ, ομοιομορφία, συγγνώμη. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση αυτό, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία και βεβαίω πάντα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τι ε, λεπτομέρειε τη πρόταση, αλλά αν υπάρχει οποιοδήποτε ερώτημα ή σχόλιο, ευχαρίστω να απαντήσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Όλσον. Ποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπουσούτιλ. Well, thank uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να αναφέρω και εγώ κάποιες αμφιβολίες που έχει η ομάδα μου με τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν τα πράγματα για το φάκελο αυτό. Κατανοούμε βέβαια και θέλουμε να τονίσουμε το υψηλό, τον υψηλό βαθμό ευαισθησίας όλων αυτών των θεμάτων που καλύπτει ο φάκελος και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να δράσουμε πολύ προσεκτικά. Ε, ασχολούμαστε με θέματα τα οποία άπτονται πολύ προσωπικών καταστάσεων των πολιτών μας και πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε πρόκληση να ρυθμίσουμε τις ζωές των πολιτών έντονα. Βεβαίως η αρχαία της μη διακριτική μεταχείρισης σημαίνει αυτό ακριβώς που λέει. Και πρέπει να την λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Είμαστε μια ομάδα που θέλει φυσικά να συνεργαστεί πλήρως για να επιτύχουμε τελικά ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό το τελικό αποτέλεσμα θέλουμε να είναι ισόρροπο αποτέλεσμα. Να μην πάει πολύ μακριά δημιουργώντας ας πούμε εξαιρετική ε, γραφειοκρατία ή ιδιαίτερο κόστος για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Με έναν τρόπο δηλαδή που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση της επικουρικότητας. Ειδικά όταν μιλούμε για τομείς που άπτονται ηθικών ε, αποχρώσεων. Αυτή είναι η γενική μου άποψη εκ μέρους του ΕΛΚ Πρόεδρε. Η συνάδελφός μου Βερονίκ Ματιό λείπει. Είναι η σκιώδη συγγήτρια για το θέμα αυτό. Και μας προτείνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, βεβαίως δηλώνοντας την πλήρη υποστήριξη για τη συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δουλεύει το μικρόφωνο μου. Ωραία. Καλωσορίζω και εγώ το γεγονό ότι ο Ραούλ είναι ο εισηγητή. Ε, πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο άνθρωπο να ασχολείται με το θέμα αυτό. Και να ευχαριστήσω επίση και την Προεδρία για την ενημέρωση του τι γίνεται στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποια κράτη-μέλη θέλουν ε, να κατακαιρματιστεί η οδηγία αυτή σε πολλές μικρότερες, γιατί θα είναι πιο εύκολα ε, θα είναι πιο εύκολο για αυτούς να την πουλήσουν, ας πούμε, στο εκλεκτικό του σώμα. Η Γερμανία είπε ότι το κόστος, ειδικά για τις αναπηρίες, θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Και μετά υπάρχει και η οδηγία για, την, ε, για το πλαίσιο για την ε, απασχόληση αλλά η Γερμανία είναι αυτή που δίνει την υποστήριξή της στο να κατακαιρματιστεί η οδηγία, ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα αναπηριών. Ρωτήτω, λοιπόν από τα κράτη-μέλη που ε, αντίκυνται, αντιτίθενται σε αυτή την οδηγία, να μας πούν γιατί ακριβώς αντιτίθενται και να είναι σαφείς. Γιατί η οδηγία αυτή τελικά επιτεύχθη πριν από πέντε χρόνια όταν αποτύχαμε να ε, επικυρώσουμε τον Μπουτιλιώνε ως ε, Επίτροπο για τα θεμελιώδη δικαιώματα τότε είχαμε πει ότι θα υπάρξει μια οριζόντια οδηγία που θα περιλαμβάνει τα πάντα. Μετά άλλαξαν άποψη, μετά από τις τέσσερις, ε, τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων και μας είπαν ότι θα υποβάλουν ε, διαφορετικές ε, οδηγίες. Το Κοινοβούλιο είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα λόγος να αντιμετωπίζεται κάποιο με διαφορετικό τρόπο σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Και γι' αυτό τώρα καταλήγουμε εδώ στην πύρινα του θέματος και για τι ε, θρησκευτικέ πεπιθήσει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων στι θρησκευτικέ πεπιθήσει, στο δικαίωμά του να πιστεύουν σε οτιδήποτε θεωρούν ότι πρέπει να πιστεύουν. Η θρησκευτική πίστη επιβάλλεται σε κάποιον. αν επιβάλλεται σε κάποιον και μειώνει το ανθρώπινο δικαίωμα αυτού του κάποιου, του οποίου του επιβάλλεται η νέα, η νέα πεποίθηση, τότε αυτό σημαίνει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλή δουλειά Πρόεδρε. Δεν έχει νόημα να λέμε σε κάποιον ότι εντάξει μπορείς να πιστεύεις ότι θέλεις αλλά δεν έχεις κανένα νομικό δικαίωμα να το, να το πιστεύεις. Δεν μπορούμε να υποβιβάζουμε την πίστη του καθενός. Πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Στον κόσμο που ζούμε δεν βασιζόμαστε πάντα στη λογική. Εγώ θα έλεγα ας διατηρήσουμε ο καθένας την πίστη τη δική του και ας, ε, ας ασπαστούμε τα όσα λέει το Ευαγγέλιο, να αγαπούμε αλλήλους. Ας δούμε τι έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για κάποιους ανθρώπους που λόγω των διαφορετικών τους πεπιθήσεων ε, εξαφανίστηκαν από προσώπου και το θέμα είναι να δούμε και πώς φερόμαστε στις ε, μειονότητές μας. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να πράξουμε το σωστό και να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τελικά την ε, συνολική αυτή οδηγία. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Η κυρία Ενετφέλντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον εισηγητή και με τον Μάικλ Κάσμαν και για τη δική μου ομάδα η οριζόντια οδηγία είναι πολύ σημαντική και πραγματικά ανησυχώ, θέλω να δω πώς, την μεταχειρίζεται το, πώς τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο και ποια είναι τα επιχειρήματα που προβάλλει. Όπως ο κύριος Μπουσούτιλ βέβαια δεν θέλω να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έξτρα κόστος, αλλά η πρακτική δείχνει ότι σε όλες τις ε, υποθέσεις που κατέληξαν τελικά σε ένα δικαστήριο, το κόστος σπάνια ήταν το πρόβλημα. Στη Γερμανία υπήρξε πρόβλημα με την εφαρμογή παλαιότερων οδηγιών. Αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που υπάρχει πολύ καλή νομοθεσία ε, που απαγορεύει την ε, διακριτική μεταχείριση έναντι αναπήρων. Το κόστος εγώ πάντα πίστευα ότι είναι το λάθος επιχείρημα για να ε, δικαιολογήσουμε την ε, διακριτική μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που είπε ο Σάιμον για το ότι θα ε, αλλάξουμε τη ζωή πολλών πάρα πολύ, θα ρυθμίσουμε τη ζωή πολλών πάρα πολύ, δεν νομίζω. αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε δικαιώματα που μέχρι τώρα δεν έχουν. Πολύ προσεκτικά βέβαια απέφυγε να αναφερθεί σε ηθικά ζητήματα, ευαίσθητα ζητήματα. Ας τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρουμε ότι πολλοί έχουν ε, πρόβλημα να δώσουν ε, τα ίσα δικαιώματα σε ανθρώπους ομοφιλόφιλους κλπ. Ας τα πούμε λοιπόν όπως πρέπει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στο οικογενειακό δίκαιο. Ε, δεν νομίζω ότι η οδηγία αυτή θα αλλάξει τα πράγματα, αλλά είμαστε υπέρ της ίσης μεταχείρισης. Παλαιότερα στην Ευρώπη το κράτος αποφάσιζε ότι αν ανήκες σε μία πιστή, αν ήσουν ας πούμε, ας πούμε καθολικός, δεν μπορούσες να παντρευτείς κάποια που ήταν προτεστάντισσα. Υπήρχαν περίοδοι στην Ευρώπη που οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να παντρευτούν κανέναν άλλον διαφορετικής πίστη. Και σε άλλα μέρη του κόσμου οι μαύροι δεν μπορούσαν να παντρευτούν λευκούς ποτέ, ποτέ δεν ανεχτήκαμε το κράτος να επεμβαίνει στις προσωπικές επιλογές του, των ανθρώπων και την επιλογή των συντρόφων τους. Γιατί λοιπόν ε, ε, ε, σε αντίθεση με όλα όσα υπάρχουν στις συνθήκες παρεμβαίνουμε τόσο πολύ σε ό,τι αφορά την επιλογή του ανθρώπου ανάλογα με τον γενετήσιο προσανατολισμό του. Γιατί, και το ίδιο κάνουμε και με την, και με την θρησκεία. Νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν συμφωνήσει, έχουν υπογράψει τις συνθήκες, τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν είναι ότι ξαφνικά το παραβλέψαμε. Οι συνθήκες υπήρχαν και σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις μεταφράσεις. Όλες οι μεταφράσεις περιείχαν τις σχετικές διατάξεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα ίσα δικαιώματα για όλους. Για όλους. Είναι θέμα αρχής. Και ελπίζω το Συμβούλιο να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη που το έχει αναλάβει η Ισπανική Προεδρία αυτό, γιατί είμαι σίγουρη πως ε, θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να υπάρξει μια οριζόντια οδηγία που να προστατεύει τα δικαιώματα όλων χωρίς καμία εξαίρεση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Ινετφέλτ. Έχω έναν κατάλογο μελών που θέλουν να λάβουν το λόγο. Ας ακούσουμε τους κιόδες καταρχήν την κυρία Μπόσκορτ και μετά τον κύριο Ντεγιάν και προτείνω να περιοριστούμε λίγο, να αυτοπεριοριστούμε λίγο στο χρόνο ομιλίας μας, γιατί υπάρχουν και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Μπόσκουρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομη εγώ. Πιστεύω από αυτά που ακούω για το τι γίνεται στο Συμβούλιο ότι υπάρχει φιλοδοξία, κάτι να γίνει και αυτό μου αρέσει. Από την άλλη μεριά, στην πράξη, βλέπω ότι τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο ρόδινα. Ακούμε τι θέλει να κάνει η Προεδρία, τι έχουν κάνει οι προηγούμενε. Κάθε φορά, όπω και τώρα, η Προεδρία λέει ότι θέλει να το ολοκληρώσει το θέμα. Και σου Σουηδική το ίδιο θέλει να κάνει. Και η Βέλγικη το ίδιο θα θέλει να κάνει. Τώρα η Ισπανία θέλει επίση να το ολοκληρώσει. Για να δούμε. Σε ποια προεδρία θα ολοκληρωθεί στην Ουγγρική. Αυτό που θέλω εγώ να ξέρω πάντως τώρα είναι η, Ισπανική Προεδρία, στην οποία έχουμε και κάθε επιτυχία, Πώ θα λύσει αυτό το γρίφο. Υπάρχουν δυσκολίε πολλέ μα τι εξηγήσανε ότι υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στις χώρε άλλες χώρες έχουν πρόβλημα με την εκπαίδευση, Άλλε χώρε έχουν πρόβλημα με την ελευθερία πεπιθήσεων. Άλλες χώρες έχουν πρόβλημα με το κόστος που απορρέει από τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας. Όντως λοιπόν πρέπει να υπάρχει 7 Ιουνίου μια πολιτική συμφωνία. Αλλά είναι πολύ περίεργη αν θα γίνει αυτό. Και έτσι για μένα αυτό το οποίο παραμένει και θέλω να μου πει και ο συγητής πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Το κείμενο είναι ένα ωραίο κείμενο, εγώ δεν θα ήθελα να αλλάξει. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις πάνω στο κείμενο της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπόσκουρτ. Ο κύριος Δεγιόμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτό που μου φαίνεται ένα θλιβερό, έτσι όπως προχωράμε με τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις είναι ότι τελικά εμείς αφαιρούμε δικαιώματα από τους πολίτες. Είπαμε ότι το Νοέμβριο κοντεύαμε σε συμφωνία, τελικά όχι. Όταν ε, υπάρχει θέμα δικαιωμάτων, τότε δικαιωμάτων των πολιτών, τότε εμφανίζονται όλα τα προβλήματα. Ενώ όταν είναι για θέματα δικαιοσύνη και τα κράτη αποφασίζουν εύκολα. Ενώ όταν πρόκειται για δικαιώματα, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε δικαιώματα στους πολίτες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη κάτι το οποίο να προσφέρει μια προστιθέμενη αξία, να είναι κάτι παραπάνω για τους πολίτες μας. Η οδηγία αυτή είναι όντω πολύ σημαντική και η Ολλανδία την έχει ζητήσει και προσέχει τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις βέβαια. Αυτό όμως που δεν δέχομαι και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι ομιλητέ το ίδιο είπαν εδώ, ότι δεν μπορεί να περιμένουμε ίσα ή να πάρει το Συμβούλιο κάποια απόφαση. Πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να υπάρξει πρόοδος σε αυτή την υπόθεση. Πράγματι κύριε Μπουσίτη, εδώ πρόκειται για την προσωπική ζωή των ανθρώπων, ανθρώπων που χρειάζονται την οδηγία αυτή για να μην υφίστανται διακρίσεις σε βάρος τους. Πρόεδρος. Ωραία. Επιστρέφω στον κατάλογο μιλητών. Ο κύριος Ιακολίνο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η οδηγία είναι ένα θέμα που αφορά τον καθένα, την κάθε οικογένεια. Όταν μιλάμε για το πώς χτίζονται τα κτίρια, όταν λέμε ε, στην αρχιτεκτονική το κτίριο να μην υπάρχουν δυσκολίες για τα άτομα με είναι επειδή αυτά επηρέουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν και τα κριτήρια τα οποία υιοθετούμε πρέπει να είναι τέτοια που να συμφιλιώνουν διαφορετικά συμφέροντα. Θυμάμαι από την αρχή που συζητούσαμε για το πρόγραμμα στη Στοκχόλμη. Εκεί υπήρχε ένα σημαντικό κομμάτι στο κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου από το Κοινοβούλιο, έχει να κάνει με τις εθνικές ευαισθησίες και με την εθνική ταυτότητα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σήμερα, σε αυτή την υπόθεση, μιλάμε για την ίση μεταχείριση προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, πληθύσεων, αναπηρίας ηλικίας κλπ. Για το θέμα των αναπηριών μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμό γυράσκει στην Ευρώπη και ίσω οδηγείται σε κάποιο είδου αναπηρία. Οπότε αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο σε βάθο. Σήμερα δεν το συζητάμε αυτό. Συζητάμε με ποιο τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και με τι πόρους μπορεί να γίνει αυτό. δεδομένων των αρχιτεκτονικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στα κτίρια. Πρέπει λοιπόν να συμβιλιώσουμε εδώ διαφορετικά συμφέροντα. Να έχουμε κοινή λογική για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπία μέσα σε μια πραγματικότητα που αφορά πάνω από 400 εκατομμύρια ανθρώπους τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους. Πρόεδρος. Υπάρχει και ένα τρίτο σκιώδη εισηγητής, συγγνώμη που δεν το είχα καταλάβει αυτό. Κύριο Κλάις, Ευχαριστώ. Ναι, όντω, είχα ζητήσει το λόγο. Δεν είμαι ιδιαίτερα σκιώδη, είχα ζητήσει το λόγο απλώ. Εν πάση εγώ θέλω να προειδοποιήσω. Προσοχή στην υπερβολική ρύθμιση και την υπερβολική γραφειοκρατία που θα αποτελέσουν μειονέκτημα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των κρατών μελών. Μην ξεχνάμε την επικουρικότητα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτή την οδηγία. Στα κράτη-μέλη υπάρχει νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε μια ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει κάτι παραπάνω. Αν, εν πάση περιπτώσει, τελικά έχουμε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, ας προσέξουμε ο αγώνας κατά των ε, διακρίσεων, που είναι απόλυτα θεμητός, να μην οδηγήσει σε έναν αγώνα κατά της ελευθερίας. Ξέρω πολύ καλά μια που φλαμαδός περί πρόκειται και ξέρω πολύ καλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ολλανδία που είναι πολύ ανησυχητικές. Μια που η αντιπολίτευση βρίσκεται στα δικαστήρια επειδή εξέφρασε κάποιες απόψεις για το Ισλάμ. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Ακούσαμε πριν για την ελευθερία θρησκείας. Ε, λοιπόν, κανένας δεν θέτει υποαφισβήτηση την ελευθερία θρησκείας. Αλλά προσοχή, οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ή δεν πιστεύουν να μπορούν να έχουν την ελευθερία να επικρίνουν άλλες θρησκείες. Το Ισλάμ για παράδειγμα που δυστυχώς δεν είναι μόνο θρησκεία αλλά και πολιτική ιδεολογία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε κύριε Σόμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως Γερμανίδα θα έχω να πω ότι έχω αντίρρηση με αυτό που ακούστηκαν για τη Γερμανία ή τέλος πάντων σε σχέση με τη Γερμανία. Όντως, στη Γερμανία υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τα θέματα και την οδηγία για την ε, διακριτική μεταχείριση. Έχει προχωρήσει τόσο μακριά στην ε, ε, Γερμανία, την, την είχε ο πράσινο συνασπισμός αναλάβει για χρόνια γιατί πραγματικά ε, υπάρχει περιορισμός των δικαιωμάτων ε, άλλων με την οδηγία αυτή. Δηλαδή ξεπέρασε πια τα έσκαμένα η οδηγία. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο μακριά πάει αυτή η αρχή της επικουρικότητας και πόσο διακυβεύεται αν προβλέψουμε εμείς πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. δεν είμαι αντίθετη με την ύπαρξη της οδηγίας για την ε, απάλληψη της διακριτικής μεταχείρισης αλίμονο, αλλά τα κράτη-μέλη δεν είναι κράτη που ε, διακρίνουν. Έχουμε την χάρτα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, ζούμε στην Ευρώπη, αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Κάθε πολίτης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, οπότε εμεί πρέπει να φροντίσουμε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από το αν είναι υγιή ή ασθενή ή οποιαδήποτε προσανατολισμό έχει στη δική του ζωή, είτε είναι θρησκευτικό είτε είναι φιλετικό, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα. Δικαιούται να έχει αυτά τα δικαιώματα. Δυνάμει και τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να μην υπερβάλλουμε, ε, να μην προσθέτουμε πάντα κάτι στην, ε, στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η γραφειοκρατία είναι δύσκολη και αυτό δεν το κατανοούν καθόλου πια οι πολίτες μας όταν φορτώνουμε συνέχεια την νομοθεσία. Οπότε ο στόχος της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί ένα αμφιβόλο πια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση της συγκεκριμένη οδηγίας. Η κυβέρνηση έχει συμπληρώσει, της Γερμανίας έχει συμπληρώσει την οδηγία με κάποιες διατάξεις, και το πλαίσιο εδώ το οποίο προβλέπεται από το ευρωπαϊκό ε, επίπεδο δεν έτυχε μεγάλης υποδοχής από την ε, Γερμανία. Αυτή η ιστορία λοιπόν ε, που προέρχεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο έτυχε κριτικής υποδοχής στη Γερμανία. Ο συνάδελφος Κάσμαν το είπε πολύ σωστά δεν είναι σωστό σε πολιτισμένες κοινωνίες να θεωρούμε ότι όλοι είναι μειονότητα. Εντάξει, μπορεί εσεί να γελάτε, αλλά αν δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τους καπνιστές εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο, ή τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ακούστηκε στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ και πώ πρέπει να περιοριστούν, να εξαφανιστούν αν είναι δυνατόν οι καπνιστέ από την Ευρώπη. Ε, και αυτοί έχουν κάποια δικαιώματα όμω. έτσι. Λοιπόν, α σκεφτούμε λίγο προσεκτικά. Δεν μπορούμε να μεταχειριζόμαστε του πάντε όπω θέλουμε. Ε, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι οι καπνιστέ είναι άρρωστοι θεωρούνται άρρωστοι. Και τι θα του μεταχειριστούμε όπω μεταχειριζόμαστε, δηλαδή τι, του αλκοολικού. Ε, Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια της συζήτησης που κάνουμε για τη διακριτική μεταχείριση. Ένα ερώτημα όμως έχω για ένα θέμα που ανέφερε η ε, εκπρόσωπος της Προεδρίας για την προσαρμογή των ιστορικών ε, κτηρίων στις ανάγκες των αναπήρων. Το, συζητούμε, το συζητούν αυτό από ό,τι είπανε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Μιλούμε για δημόσια κτίρια ή για τα πάντα, για όλα τα ιστορικά κτίρια Δηλαδή ένας άνθρωπος με αναπηρία πρέπει να έχει το δικαίωμα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε, οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο, σε οποιοδήποτε κτίριο. Στη Γερμανία αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί ακόμη δεν, και λόγω των ε, περιβαλλοντικών αλλαγών δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ε, δυνατότητα ε, το χτίσιμο των, κτίριων. κτηρίων. Οπότε αυτό πρέπει να μα πείτε τι ακριβώ εννοείται στο, στην πρόσβαση των αναπήρων, στα, στους χώρου όλα τα κτίρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα απλώς να θυμίσω εδώ στα μέλη ότι σήμερα συζητούμε το, το σχέδιο οδηγίας ε, του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση των ανθρώπων. Είναι θέμα και ηθικό και πολιτικό. Δεν είναι τεχνικό. Αυτό νομίζουν κάποιοι, ότι είναι τεχνικό το θέμα. Δεν μιλούμε για κτίρια. Δεν μιλούμε για αρχιτεκτονική. Μιλούμε για ανθρώπους. Ανθρώπους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό καταρχήν είναι θεμελιώδες. Μιλούμε για ανθρώπους και το πώς κατανοούμε τους ανθρώπους. Η οδηγία που μας έχει υποβάλει η Προεδρία και αυτά που μας είπε η εκπρόσωπος της Προεδρίας, φαίνεται ότι τη χάνει και αντίθετων απόψεων και, στην, και στο Συμβούλιο. Πρέπει να θυμόμαστε όμως και εμείς εδώ, να μην μετατρέψουμε το θέμα αυτό που είναι βαθιά ηθικό σε ένα τεχνικό θέμα. Μιλούμε για το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ποιον, με ποιον ζουν, πώς θα ζήσουν τη ζωή τους, ποια μεταχείριση θα τη χάνουν, αν θα πρέπει να την χάνουν ίσε μεταχείριση ανεξάρτητα από το αν έχουν αναπηρία ή όχι. Αυτά είναι δεδομένα, δεν θα έπρεπε να τα συζητούμε. Λυπάμαι τώρα που θυμώνω τόσο πολύ, αλλά είμαστε στον 21ο αιώνα, Πρόεδρε. Μιλούμε για δικαιώματα, δεν μιλούμε ούτε για τη θρησκεία, ούτε για το δικαίωμα τη θρησκεία. Αυτά είναι δεδομένα πράγματα. Μιλούμε για την ελευθερία τη επιλογή θρησκεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ίσως να είμαι η μόνη σε, αυτό το, σε αυτή την αίθουσα σήμερα που είμαι και ιερέας και έχω έτσι μια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Πραγματικά με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ που αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα μετατρέπεται σε μια τεχνική λεπτομέρεια, σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Όταν μιλούμε για την πρόσβαση, α πούμε, στα κτίρια δεν, δεν αξίζει η Επιτροπή αυτή να, υπο, να μετατρέπει αυτό το πρόβλημα σε, σε μια λεπτομέρεια. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πολεμούμε, για να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη ζωή τους και να την ζουν όπως θέλουν. Δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης αυτό. Προσπαθούμε να εδραιώσουμε το, το δικαίωμα κάποιου να είναι άνθρωπο το 2010 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2010 και να εδρεώσουμε τι ελευθερίε που έχει. Μα είναι δεδομένε αυτέ και μπορεί να τι επιλέξει και μπορεί να επιλέξει με ποιον θα ζήσει, πού θα ζήσει και πώ θα ζήσει. Αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κρατημέλη παντού και πάντα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον εισηγητή ότι ελπίζω να μπορέσει με ενθουσιασμό και με ζήλο να εργαστεί για την έκθεσή του. Ελπίζω και η Ισπανική Προεδρία να μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να προχωρήσει. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά ανθρώπους, ανθρώπινα όντα. Για σας, για μένα, για όλους τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημασία αυτό. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2010 πρέπει κάποιος να έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να διαλέγει πώς θα ζήσει, πού και με ποιον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόγκς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να να μην υπάρχει ε, άδικη μεταχείριση των ε, εργοδοτών έναντι των εργαζομένων. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες χωρίς να υπάρχει λόγος. Μιλούμε για θρησκείες, για δόγματα, ε, ποιον θα έχει δικαίωμα κάποιος να θέσει ως ιερέα. Επίσης, τα πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να, στα πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να λέμε πώς θα ασκήσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες ή ποιες θα είναι οι πολιτικές τους ε, πεπιθήσεις. Δεν προωθούμε έτσι την ελευθερία, αλλά βάζουμε περιορισμούς και στις πολιτικές ελευθερίες και στις θρησκευτικέ ελευθερίες. Φαίνεται ότι οι θρησκευτικέ και οι πολιτικέ ελευθερίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι εξαρτώνται από τα πολιτικά κόμματα που ε, υπογράφουν τις ε, ε, αρχές αυτές του φιλελευθερισμού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τελειώσαμε νομίζω. Βλέπω και κάποιον άλλον. Βλέπω και κάποιον άλλον που θέλει το λόγο για να δώσουμε μετά το λόγο το Συμβούλιο και να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Κροτσέλα το λόγο. Πρόεδρε, εγώ άκουσα πολλές τοποθετήσεις για πολλές πλευρές. Και κάποιος αναφέρθηκε στην ελευθερία του θρησκεύματος. Μα αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα σήμερα στην Ευρώπη. Διότι αν εμείς ε, αναλογιστούμε τι, γίνεται, τι έγινε στην ε, Ελβετία με το δημοψήφισμα για τους μιναρέδες, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έγκαιρα ότι μέσα στην ίδια την Ευρώπη θα μπορεί να γεννηθούν κινήματα τα οποία είναι εθνοφοβικά, όπου θα, αρνούνται την συνύπαρξη των διαφόρων θρησκειών. Ας πούμε η συζήτηση για τους μιναρέδες ε, ε, έγινε στην Ελβετία η σύγκριση σαν συγκρίνοντας τους ε, μιναρέδες με τους πυράβλους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα ατομικά ε, δικαιώματα για τις ε, ατομικές ελευθερίες αλλά επίσης και τα συλλογικά δικαιώματα άσκησης ε, θρησκείας διότι αυτό είναι μήμα του κράτους των εγγύσεων που παρέχει το κράτος δικαίου και όπου τα δικαιώματα δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα ε, σημεία για συζήτηση. Σας παρακαλώ, όποιος θέλει να πάρει το λόγο, ας είστε σύντομοι. Σοφή. Πρόεδρε, κάτι που είπε η κυρία Σόμερ ήθελα να σχολιάσω. Γιατί αναφερθήκατε στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και γιατί χρειαζόμαστε ε, οδηγία, αφού υπάρχει η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που του δίνει την προστασία την απαιτούμενη. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λέτε αυτό. Όταν συζητούμε εδώ σε πολλέ περιπτώσει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε κάποια κράτη-μέλη σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης ή μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ΕΛΚ ήταν αυτό που είπε ναι αλλά η χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις συγκεκριμένες εξουσίες. Οπότε, αν δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι συγκεκριμένε εξουσίε, πώ δίνει εξουσίε στου μεμονωμένου πολίτε. Τι ακριβώ εννοεί το ΕΛΚ όταν το λέει αυτό. Ας μην ξαναρχίσουμε όμως τη συζήτηση, Σόφη, τώρα. Κύριε Μπουσούτιλ, εντάξει, θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Κάσμαν, όχι. Ωραία. Ο κύριος Μπουσούτιλ και μετά στον κύριο Ρωμέβα ο λόγος και στην Προεδρία. Πρόεδρε, δυστυχώς, εδώ έχει λάθος εντύπωση ότι αν δεν ακολουθήσει κανείς τη γραμμή της Σόφη ή της κυρίας Βίκμαν πιο πριν ε, στις παρεμβάσεις της, τότε είναι κανείς αντίθετος στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, απλώς έχουμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές πολιτικές απόψεις και απλώς θέλω να τις σεβαστείτε, να σεβαστείτε τη διαφορετική μας άποψη. Αυτό που ήθελα εγώ να πω και σε σχέση με αυτό που είπε η Σόφη είναι το εξή. Αυτό που λέμε εδώ δεν είναι ότι είμαστε αντίθετοι με τους ανθρώπους, με τους πολίτες μας, όπως είπε η κυρία Βίκμαν, ή ότι είμαστε αντίθετοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε άλλο παρά. Είμαστε υπέρ της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης. Μάικολ, πίστεψέ με, είμαστε υπέρ της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν και όρια στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πόσο μακριά μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετώντας επί τη βάση της αρχής της επικουρικότητας. Για αυτή την αρχή, αυτή η αρχή είναι αυτή που θα έπρεπε να γίνεται σεβαστή. Δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε, να τη διαγράψουμε. Είναι τμήμα των συνθήκων. Αυτό είπαμε απλώς. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, δύο δευτερόλεπτα. Εντάξει, δεν θα απαντήσουμε στα πάντα εδώ, αλλά αν το ΕΛΚ θεωρεί ότι η Χάρτα των Θεμελιών Δικαιωμάτων δεν δίνει εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει ε, τα δικαιώματα των πολιτών της στα κράτη-μέλη, πώς δίνει εξουσίες στους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η συζήτηση ε, ξανανοίγει, ξανακλίνει, ξανανοίγει. Ε, ας τελειώσουμε κάποια στιγμή γιατί ο κύριος Κάσμαν ε, μας είπε να διατυμπανίσουμε κι εμείς το, το Ευαγγέλιο, να αγαπάμε αλλήλους. Εδώ δεν φαίνεται να αγαπάμε πολύ αλλήλους τώρα με τη συζήτηση, ας καταλήξουμε κάπου. Μια ανταλλαγή απόψεων κάνουμε. Εντάξει, μην συγχυζόμαστε τώρα τόσο πολύ. Κύριε Σόμερ. Δεν θέλω να ξαναξεκινήσουμε, Πρόεδρε, μια τέρμονη συζήτηση. Απλώς είπα ότι δεν μπορεί να απαντήσει κανείς πάντα έτσι άμεσα σε αυτά που ακούει. Εγώ απλώς ε, ήθελα να... Ε, μου είπατε ότι προσπαθώ να σας ε, κάνω μάθημα. Ε, κυρία συνάδελφε, περιμένετε, μιλάω εγώ τώρα. Ε, μόλις σηκώστε το χέρι σας, θα λάβετε τον λόγο, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, υπάρχει χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτά πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Ως εκεί συμφωνούμε. Το έχουμε χαιρετήσει, έχουμε την συνταγματική συνθήκη, έχουμε τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είμαστε μέλη, έχουμε τη συνθήκη τώρα της Λισαβόνας. Θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε ε, ότι μάλλον θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν και διαφορετικέ απόψει, οι οποίε όμω εξακολουθούν να είναι υπέρ της, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα είναι μέχρι πού θέλουμε να πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά είναι σωστό να εμπλεκόμαστε, να συμμετέχουμε όταν ας πούμε κάτι σε ένα κράτος μέλος δεν πάει καλά, όταν υπάρχει παραβίαση θεομελιωδών δικαιωμάτων και αυτό αναφέρεται και στη συνταγματική Συνδίκη και, και στη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά το θέμα είναι μέχρι πού η επιπλέον νομοθεσία πρέπει να προχωρήσει. Εμείς είμαστε υπέρ να έχουν όλοι να την χάνουν όλοι ίσει μεταχείριση, να μην υπάρχει διάκριση κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε. Α μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία υπάρχουν 27 κράτη-μέλη, 27 δημοκρατίες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν, ε, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει τίποτα στα κράτη αυτά. Εγώ δεν είπα τίποτα από αυτά που είπατε εσείς, ε, κυρία Ινετφέλντ. Εντάξει. Ο κύριος Κάσμαν. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πρόθεση του Κοινοβουλίου, κάπου 11 χρόνια με εδώ, είναι να φροντίζει, να δικατοπτρίζει ακριβώς αυτά τα οποία αναφέρονται στην οδηγία για τον ρατσισμό κτλ. Φυσικά και υπάρχει επικουρικότητα και γι' αυτό και το ΕΛΚ πρέπει να αναγνωρίσει τα θετικά της οδηγίας αυτής. Θα είναι μεγάλη πρόοδος. Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επικουρικότητα. Γιατί εμεί λέμε ότι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία χώρα είναι το ίδιο σαν να πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων στη δικιά μου τη χώρα. Και γι' αυτό συνυπογράψαμε την Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Ο κύριο Κορτσέτα ακόμα. Σύντομα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει εμείς να προσεγγίζουμε μέσα από την αρχή της ανοχής τα δικαιώματα. Ανεχόμαστε κάποιον γιατί είναι διαφορετικός από σένα, γιατί πρέπει να τον κανακεύεις, να τον προσέχεις, σαν να είναι δηλαδή κάποιος ε, δεύτερης κατηγορίας. Εμείς εδώ να αφήσουμε ήσυχη την αρχή της επικουρικότητας και πρέπει να πούμε ότι είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρει όλα εκείνα τα εμπόδια τα οποία υφίστανται στην κράτη-μέλη και εμποδίζουν την απόλυτη ισότητα μεταξύ των πολιτών. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι για να καταλήξουμε πρώτα ο εισηγητής και μετά η Ισπανική Προεδρία. για ο κύριο Κάσμαν είναι εισηγητής για το επόμενο θέμα μα και πρέπει να φύγει γύρω στι 5. Οπότε πρώτα ο κύριο Δομεύο και μετά η Ισπανική Προεδρία γρήγορα παρακαλώ. Ας προσπαθήσουμε να μην επανεφεύρουμε τον τροχό. Είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε καταλήξει σε ένα συνενετικό κείμενο και ζήτησα μάλιστα και από τη γραμματεία να το μοιράσω σε όλους τους συναδέλφους για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Θα μας βοηθούσε να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και περί τίνος δεν πρόκειται. Δεύτερον, ως εισηγητής θα ήθελα παρόλα αυτά να υπογραμμίσω ότι η σειρά μπορεί να είναι και διαφορετική της προσέγγισής μας. Δηλαδή, αντί να ξεκινάμε από το κόστος, εγώ προτιμάω να μιλάμε για το ωφέλη, τα κοινωνικά ωφέλη από την μη διάκριση. Φυσικά και έχουν γίνει συζητήσεις για το κόστος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το κόστος αυτό όμως αντισταθμίζεται κατά πολύ από τα κοινωνικά ωφέλη που προσφέρει η μη διάκριση σε ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι πρέπει να το δούμε. Γι' αυτό και να χρησιμοποιούμε τους σωστούς όρους, τη σωστή διατύπωση. Τώρα, για το θέμα της συνοχής ή όχι. Πώς όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ως επιπλέον νομοθεσία. Τώρα δημιουργούνται αμφιβολίες. Γιατί λέμε ότι στο ένα κράτος μπορεί κανείς να τυχαίνει διάκριση για ένα λόγο και σε μια άλλη χώρα όχι. Ε, αυτό είναι που πρέπει να λυθεί. Και πρέπει να λυθεί και γρήγορα. Δεν μπορεί στη μια χώρα να θεωρείται κάτι διάκριση και σε μια άλλη όχι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τέλος. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Πολλά πρέπει να λυθούν γρήγορα και αυτό που θέλω να ζητήσω από το Συμβούλιο και να ρωτήσω εμείς πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και εσείς πώς σκοπεύετε να ζητήσετε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις συζητήσεις. Δεδομένου ότι ο ρόλος που μπορούμε να παίξουμε στις συζητήσεις αυτές θα βασίζεται στη συμφωνία που θα έχει προηγουμένως ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε η Ισπανική Προεδρία τώρα για να καταλήξει για αυτό το θέμα, να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους μίλησαν, όλους τους βουλευτές και βουλευτίνες, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σημειώσαμε όλα όσα μας είπανε. Και θέλω να επαναλάβω ότι οι εργασίες αυτή την οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι μια οδηγία πολύ σημαντική, πολύπλοκη και η δουλειά μας είναι σοβαρή και ιδιαίτερα προσεκτική. Και συνεχίζει η Ισπανική Προεδρία και την δουλειά των προκατόχων της. Θα καταβάλουμε λοιπόν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε καλύτερα τις διαπραγματεύσεις. Είναι θέματα πολύπλοκα, απαιτούν χρόνο διαπραγματεύσεις, ορισμούς ε, ε των διαφόρων ενιών, καθορισμό των ενιών αυτών. Η κυρία Ζόμερ ε, ρώτησε για τα ιστορικά κτίρια. Εγώ τώρα παράδειγμα σας έδινα για τη δυσκολία που θέτει η οδηγία, που είναι μια δύσκολη οδηγία. Επίσης χρειάζεται ομοφωνία μετά από την έγκριση από το Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η δυσκολία σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ. Ευχαριστούμε την Ισπανική Προεδρία. Ακούσαμε τι η Επιτροπή θέλει να αντιδράσει. Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί από την Ισπανική Προεδρία και την δέσμευσή της πάνω σε αυτό το θέμα. Τους ευχαριστούμε. Τώρα προς τον εισηγητή και για τα σχόλια που έγιναν. Η οδηγία αυτή δεν προσπαθεί να διακανονίσει τα πάντα στην κοινωνία. Πρόκειται για την πρόσβαση σε αγαθά. Αυτή είναι η συζήτηση. Μην μπαίνουμε λοιπόν τώρα σε άλλα παράπλευρα θέματα. Είναι σημαντικά και αυτά, αλλά δεν θα λυθούν με αυτή την οδηγία. Το άλλο, για την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες, όπως είπε και ο συγητής, έχει κοινωνικά θετικά, κοινωνικά πλεονεκτήματα, αλλά και οικονομικά. Γιατί όσοι δεν έχουν πρόσβαση στα αγαθά ή στις υπηρεσίες, δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Και αυτό είναι κόστος για την ε, οικονομία μας. Ευχαριστούμε, ωραία. Και έτσι εδώ κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα, προς το παρόν βέβαια. Γιατί η συζήτηση ξεσηκώνει τα πάθη. Αλλά ο χρόνος περνάει και πρέπει να περάσουμε γρήγορα στο επόμενο θέμα που είναι πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Με εισηγητή τον κύριο Κάσμαν. Προτείνω χωρίς άλλη να του δώσουμε το λόγο. Ενημερώστε μας για την κατάσταση πραγμάτων. Η ανταλλαγή απόψεων θα λάβει χώρα αμέσως μετά την παρουσίαση του εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι πράγματι σύντομος γιατί αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μέχρι σήμερα. Μετά το ψήφισμα που είχαμε στην Ολομέλεια, νομίζω ότι τώρα, επειδή είμαστε σε πρώτη ανάγνωση ακόμα, έχουμε την ενημερωμένη πρόταση της Επιτροπής, που δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλά σίγουρα προσαρμόστηκε κάπως και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό που θα ήθελα εγώ τώρα να κάνω τις επόμενες μέρες είναι να ετοιμάσω ένα σχέδιο έκθεσης. Σε αυτό το στάδιο και δεδομένων των συζητήσεων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συνολική συμφωνία, τέλος πάντων να ξεκινήσω με μια πρώτη θέση βάσει της τοποθέτησης του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2009. Και αυτό από κοινού με την νομική υπηρεσία που θα γνωμοδοτήσει βάσει της νέας συνθήκης. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου καταρχήν. Και μετά στην Ολομέλεια να έχουμε μια πρώτη ανάγνωση εφόσον έχει γίνει η συζήτηση και η ψηφοφορία στην δικιά μας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ελπίζω να συμφωνήσουν και οι σκιώδες εισηγητές. Έχω εδώ πέρα ένα σημείο μου, η κυρία Χάουταλα, επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Προβλέθηκε συζήτηση και με εθνικούς βουλευτές. Δεν μπόρεσαν να έρθουν όμως. Αλλά έτσι καλώς δεν έχουμε χρόνο, οπότε μάλλον τόσο το καλύτερο. Θέλω να ακούσω τους σκιώδες εισηγητέ και την Επιτροπή τι έχουν να πούνε. Αν και η Επιτροπή υποθέτω ότι δεν θα έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσθέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν που μας ενημερώσατε και τόσο γρήγορα. Εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κύριος Κρίστινσεν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή χαίρεται για το κείμενο του, Επιτρο... του Κοινοβουλίου και τη θέση του του Δεκεμβρίου. Επιβεβαιώνουμε αυτά που είπε ο κ. Κάσιμαν, ότι δηλαδή θέλουμε το Κοινοβούλιο πράγματι να προχωρήσει και να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση βάσει της συνηθισμένη θεσμική πρακτικής. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε στη διαδικασία όπου τα τρία θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να έχουν καρποφόρο διάλογο και να οδηγηθούν σε ό,τι τροποποίησης χρειάζεται πολύ σύντομα. Η κυρία Μπενίτο τώρα, Ισπανική Προεδρία, θέλετε το λόγο? Κυρία Μπενίτο, θέλετε το λόγο? Όχι? Καλώς. Οι ευρωβουλευτές τότε. Η κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό. Έχουμε συζητήσει αρκετέ φορέ και στην Ολομέλεια, αλλά έτσι γίνεται στις ε, δημοκρατίες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της αποψή του. γεγονό είναι, και το είπε και ο εισηγητή και έχει δίκιο, ότι αυτός ο φάκελος ε, εκρεμεί εδώ και καιρό. Από την τελευταία, από την προηγούμενη θητεία μάλιστα. Ε, και κάποια στιγμή κάπω πρέπει να προχωρήσουμε ε, με το ψήφισμα εγώ, η δική μου ομάδα δεν συμφωνούσε. Εν πάση περιπτώσει πέρασε στην Ολομέλεια. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με το φάκελο αυτό. Δεν γίνεται να ξανακρατήσει άλλα πέντε χρόνια και να μείνει στα σιρτάρια μας. Εγώ ευχαρίστω να έρθω σε επαφή και με τους σκιώδεις και με τον εισηγητή, να ανταλλάξουμε απόψει. Ε, ίσως καλό θα ήταν και εκ μέρους της Κομισιόν αν και είπε η την τη Κομισιόν, ε, δεν ακούσαμε πάρα πολλά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσω να έρθουν οι σκιώδει σε επαφή με την Κομισιόν, γιατί ε, ξαναξεκινά η διαδικασία, έχουμε και τα είναι Λισαβόνα, οπότε ίσως να υπάρχουν νέες εν τω μεταξύ πληροφορίες. Εγώ ευχαρίστω να συμβάλλω, να βοηθήσω για να προχωρήσουμε μπροστά με το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. No more comments. Wow, Κύριε Κάσμαν, τα καταφέρατε. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω στις 5, γιατί θα μιλήσω απόψε μετά τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας για την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση. Οπότε θα τον ενημερώσω και για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σόμερ για τα σχόλιά της και για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το φάκελο. Δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά ε, έτσι πρέπει να προχωρούμε στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που να καλύπτει όλα τα μέρη. Ο κύριος Διόν που είναι εδώ Επίσης υπήρξε πολύ επικοδομητικός, μας βοήθησε πάρα πολύ για να προχωρήσει ο φάκελος. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο, πέρα από το γεγονός ότι θα έλεγα στους αγαπημένους φίλους της Κομισιόν ότι ε, δεν γίνεται πάντα να μας βάζετε στην γωνία και να μας κατηγορείτε ότι δεν κάνουμε καμία πρόοδο επειδή δεν ακολουθούμε τη συνήθι θεσμική πρακτική ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ανάγνωση. Στο 90% ε, των φακέλων της συναπόφασης πριν τη Λισαβόνα αυτής της Επιτροπής πάντα κατέληγαν σε συμφωνία. Πριν την ολοκλήρωση ή πριν ε, γίνει η ε, πρώτη ανάγνωση. Απλώς για το τυπικό το λέω αυτό, γιατί αυτό το να μας κατηγορούν συνέχεια μάλλον πίσω μας πάει και όχι μπροστά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Τώρα θα προχωρήσουμε στην πρώτη ανάγνωση, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ποιο, ναι, ο κύριο Μπουσούτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη, μήπω μπορώ να ρωτήσω, μήπω μπορώ να ζητήσω να αναβάλουμε το σημείο 9 για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια από. Ε, ο εισηγητή δεν είναι εδώ. Η εισηγήτρια, συγγνώμη, δεν είναι εδώ. Και ξέρω ότι και πολλά ε, μέλη πρέπει να φύγουν, να τρέξουν στα αεροδρόμια. Οπότε, μήπω θα μπορούσαμε να το αναβάλουμε για μια επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Βεβαίω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα, θα το αναβάλουμε. Θα το συζητήσουμε σε μια μεταγενέστερη συνεδρίαση. Οπότε, μια που, αν θυμάστε, ακυρώσαμε το 7 για τη διαρευνητική αποστολή στο νότιο τμήμα της Ιταλίας, πάμε στο 8. Σωστά τα λέω. Ε, το Και το 8 έχει διαγραφεί. Α, οπότε το επιπλέον σημείο για την ε, παρουσίαση από την Επιτροπή ε, έγινε. Ο κύριος Φόλ ήταν εδώ. Το σημείο 8 λοιπόν ολοκληρώθηκε. Το 9 το αναβάλαμε. Οπότε κλείνουμε για σήμερα. Καλό σας απόγευμα.